to ψήφου. Για την έκθεση Τσβέρ, ο κύριος Γιακολίνος. Ναι κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συγκεκριμένη έκθεση αποτελεί ένα βήμα προς το μέλλον για τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων επιμόρφωσης ε, των νέων με περισσότερη έρευνα, καλύτερη στρατηγική για το 2020 σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι όλο ένα και πιο επίκαιρο πιο ε, σχολική παιδεία, πιο κατάρτιση αλλά και περισσότερη ε, πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Αυτό θα μπορέσει να συνεισφέρει λοιπόν στους νέους οι οποίοι αποτελούν και προστιθέμενη αξία για την προαγωγή του πολιτισμού να υπάρχει μια δυνατότητα επιμόρφωσης. Ε, είναι αυτό το οποίο προωθεί η έκθεση και γι' αυτό και υπερψηφίσαμε. Ζητούμε περισσότερη κινητικότητα για τους νέους, μεγαλύτερες δυνατότητες ε, το ανάπτυξης των ευκαιριών εργασίας, εργασία η οποία δεν θα πρέπει να βλέπει μόνο τους νέους αλλά και όλους όσους ε, έχουν δυνατότητα ανάπτυξης όπως και οι νέοι. Ο κύριος Κόσλικ. Frau Präsidentin! Mr. Koslick. Frau Präsidentin, geht nicht. No micro. No, it's for Mr. Koslick, not you, Mr. Posselt. Όχι για σας κύριε Πόσελτ. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι βουλευτές, εγώ υποστήριξα την πρωτοβουλία Youth on the Move που στοχεύει στη μείωση των εγκαταλείψεων από το σχολείο μέχρι το 2020 από το 15% στο 10% και στην αύξηση της αποφύτησης στο 40% ε, τουλάχιστον. Στην Ιαπωνία όμως οι επιτυχίες φτάνουν το 50%. Μέχρι σήμερα οι νέοι από 18 μέχρι 24 μόνο κατά 18% πηγαίνουν σε ανώταρη εκπαίδευση και παραμένουν οι περισσότεροι άνεργοι. Γι' αυτό ετάχθην υπέρ της πρωτοβουλίας αυτής Youth on the Move. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 20 θα υπάρχουν περισσότερες ανάγκες για πανεπιστημιακά διπλώματα. Κολινόφσκι. Καλινόφσκι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευρωπαϊκά προγράμματα που υποστηρίζουν την νεολαία χρειάζονται την υποστήριξή μας. Γιατί εδώ μιλάμε για το μέλλον μας, για το μέλλον της Υπήρου μας και η νεολαία βρίσκεται σε πολύ ευάλωτη θέση σήμερα. Πρέπει να μάθει γλώσσες, πρέπει να επιμορφωθεί επαγγελματικός για να έχει αληθινά επιλογή. Δεν μπορούν όλοι να πληρώσουν τέτοια παιδεία μόνοι τους. Υπάρχουν τα προγράμματα Έρασμος και Λεωνάρδος, αλλά και έχουν αποδείξει την αξία τους. Ιδιαίτερα οι νέοι από την Ήπεθρο έχουν λιγότερες ευκαιρίες να παρακολουθήσουν ανώτερη εκπαίδευση. Τάκουλας. Κυρία Πρόεδρε, για την κάλλιστη αυτή έκθεση Youth on the Move θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για μία από τις λίγες επιτυχημένες ιστορίες που μπορεί να μας διηγηθεί η Ένωση. Ακόμα και οι ευρωσκεπτικιστές και ευρωσκεπτικίστριες συμφωνούν ότι η δυνατότητα που πρέπει να δοθεί στους νέους ιδιαίτερα της υπαίθρου είναι κάτι το θετικό. Γι' αυτό η έκθεση του κυρίου Τσβέρ ενδυναμώνει τις θετικές τάσεις που συμφωνούμε ότι υπάρχουν στην κοινωνία μας γιατί δίνει περισσότερες ευκαιρίες στους νέους για να σπουδάσουν σε άλλες από τη δική τους χώρες. Και μακροπρόθεσμα πιστεύω ότι θα είναι από τις ισχυρότερες βάσεις για την μελλοντική μας οικονομική ανάπτυξη και ακόμη παραπάνω θα δώσει τη δυνατότητα σε μεγαλύτερη ανθρώπινη ανάπτυξή τους, εξέλιξή τους. Πρόεδρε, εδώ σε ολόκληρη την Ευρώπη καταδικάζουμε ολόκληρες γενιές στην αποδημία και στην ανέχεια, ακόμη και στους αγενήτους. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε πια αυτήν την απάτη όταν ξέρουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν συνεχώς εξεγέρσεις κατά των μέτρων λιτότητας, στην Ιρλανδία ξέρουμε τι συμβαίνει και γνωρίζουμε ότι όλα αυτά δεν φέρουν αποτέλεσμα, τα μέτρα δηλαδή ότι θα είναι προσωρινά και δευτερεύοντα μέτρα βλέπουμε ότι έχουν ήδη αποτύχει και συνεχίζουμε παρόλα αυτά την ίδια πολιτική και στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα ξανά πρέπει να παραδεχτούμε το λάθος μας και την ψηλή τιμή που περιμένουμε να πληρώσουν οι φορολογούμενοι μας η κυρία Σμολκονάιτε Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί σήμερα εγκρίναμε τις προτάσεις Youth on the Move η οποία κάνει σαφείς συστάσεις ως βάση για την προώθηση της καλύτερης εκπαίδευσης της νεολαίας. Καταρχήν η πρωτοβουλία Youth on the Move στοχεύει το 2020 να μειωθεί ο αριθμός των εγκαταλειπώντων τα σχολεία από το 15% στο 10%. Και στη βελτίωση των προσόντων και των διδασκόντων οι οποίοι αντιμετωπίζουν και αυτοί προβλήματα. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι Ευρωπαίοι διδάσκαλοι θα είναι οι καλύτεροι του κόσμου. Χαιρόμαστε γιατί η Κομισιόν συμφωνεί να υπάρξει μια σφαιρική στρατηγική για την παιδεία. Ε, σας ευχαριστώ ιδιαίτερος γι' αυτό. Ο κύριος Πόσελτ, κύριε, Πρόεδρε, είμαι και μέλος της οργάνωσης ε, της νεολαίας των Σουδητών και προωθούμε τη συνεργασία με την τσεχική νεολαία. Η έκθεση λοιπόν για μας έχει τεράστια σημασία διότι περιλαμβάνει τρεις παραγράφους. Την διαδικτύωση των πανεπιστημίων ιδίως στις ευρωπαϊκές περιφέρειες και παραμεθόριες περιφέρειες, την επαγγελματική κατάρτιση διότι δεν αρκεί βέβαια μόνο η πανεπιστημιακή και η εκμάθηση γλωσσών. Κυρία Πρόεδρε, λατρεύω την γλώσσα του Σέξπιρ αλλά βρίσκω κρίμα οι νέοι να μιλούν και να συνεννούνται μεταξύ τους μοναχά σε μία γλώσσα καλύτερα να μάθουν και τη γλώσσα του γείτονα. Πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε ιδίω αυτέ τι γλώσσε, διότι μόνο έτσι γνωρίζει κανεί πραγματικά και τον πολιτισμό του γείτονα όταν αρχίσει να μαθαίνει και να κατέχει καλά τη γλώσσα του. Thank you, Mrs. Mrs. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που η πρωτοβουλία νεωρέα εκκίνηση αποτελεί μέρος της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Μιλούμε για εκπαίδευση και επίσημη και ανεπίσημη, για συνεργασία με οργανώσεις νέων, μη κρατικές οργανώσεις. Εγώ θεωρώ ότι η εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει τους νέους να αναπτύξουν την κοινωνικοποίησή τους και να έχουν περισσότερες εν τέλει πιθανότητες να απασχοληθούν στην αγορά εργασίας. Έκθεση Hannibal για την μάθηση στα νερά χρόνια της ηλικία Καλινόφσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για το μέλλον των παιδιών που στις προσπάθειές τους θα βασιστεί η νέα κοινωνία και γι' αυτό χρειάζεται να εκπαιδεύονται τα παιδιά από την τρυφερή ηλικία. Η εκπαίδευση πρέπει να βασιστεί σε γερά θεμέλια και να γίνεται βεβαίως από καλά καταρτισμένους δασκάλους. Χρειάζεται επίση να εξασφαλίσουμε ίσους όρου ανταγωνισμού για όλα τα παιδιά από όπου και αν προέρχονται πόλεις, χωριά, φτωχότερε φτωχότερες περιφέρειες. Όλα τα παιδιά πρέπει να χαίρουν των ίδιων ευκαιριών, να έχουν ίσες ευκαιρίες στη ζωή του. Και κυρίως παιδιά από αγροτικές περιφέρειες πρέπει να έχουν περισσότερες ικανότητες να μπορέσουν να φτάσουν στα πανεπιστήμια. Τάκουλα για την έκθεση Hannibal. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικό να ρίξουμε ιδιαίτερο βάρος στην ε, μάθηση από την παιδική ηλικία. Η έκθεση είναι καλή, αλλά θα ήθελα παρόλα αυτά ε, να συνοδεύεται και από το εξή. Η εκπαίδευση από νεαρή ηλικία των παιδιών. Θα δώσει τα θεμέλια στα παιδιά. Το παιδί χρειάζεται ασφαλές περιβάλλον για να μπορέσει να αναπτυχθεί και αυτό είναι σημαντικό γιατί έτσι θα μπορέσει να αναπτύξει την προσωπικότητά του και για το μέλλον. Άρα εκπαίδευση, σχολική εκπαίδευση είναι σημαντικά πράγματα και αυτά τα γράφει καθαρά η έκθεση. Υπάρχουν διάφορα πρότυπα στις διάφορε χώρε μέλη, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να φροντίσουμε ώστε κανένα παιδί στην Ευρώπη να μην στερείται της δυνατότητας να προχωρήσει στην εκπαίδευσή του. Μία φορά πήρα τα παιδιά μου στην παραλία και είδα τις δύο κορούλες μου να φτιάχνουν ένα κάστρο στην άμμο χωρίς να προσέχουν τα ε, κύματα που σιγά σιγά και να το στολίζουν. Εγώ δεν είχα, το, δεν είχα τη διάθεση να τους πω προσέξτε θα χάσετε το κάστρο σας γιατί έρχονται τα κύματα. Το ίδιο έχουμε και σήμερα την κατάρρευση του ε, ακαθάριση του εθνικού προϊόντο μα Μιλούμε για εκπαίδευση, κατάρτιση για το μέλλον, για το Σαράγεβο να είναι πολιτιστική πρωτεύουσα τη Ευρώπη, Αλλά ποιε είναι οι στατιστικέ. Το 1974 οι χώρε τη Δυτική Ευρώπη είχαν το 36% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Για το 2020 θα είναι το 15%. Όλα λέμε αυτά τώρα προπαγάνδα για μικρή ηλικία και εκπαίδευση Όλα αυτά είναι γελία διότι ε, υπάρχουν άλλες χώρες πολύ πιο ε, ρωμαλαίες αυτή τη στιγμή που έχουν διδαχθεί σωστά τα διδάγματα της αποκέντρωσης. Μήπως εκεί πρέπει να στραφούμε κι εμείς. Και αμόκινάεται. Θα ήθελα να απαντήσω στη συζήτηση και στην δήλωση του ε, Ευρωβουλευτού Τομασεύσκη που δεν είναι αληθινή, δεν είναι ορθή ότι τα οι νεαροί Πολωνοί στην Λιθουανία δεν μπορούν να διδαχθούν την ε, ε, πολωνική γλώσσα. Όχι, υπάρχουν σχολεία που τους προσφέρουν την εκπαίδευση σε πολωνική γλώσσα. Ενώ στη Γερμανία με πολύ σημαντικότερο αριθμό Πολωνών ε, μεταναστών δεν υπάρχει ε, τέτοια δυνατότητα. Στη Λιθωνία τα παιδιά των Πολωνών διαθέτουν εκπαίδευση σε πολωνική γλώσσα από τον ε, παιδικό σταθμό μέχρι το πανεπιστήμιο. 42% των εθνικών μειονοτήτων στην Λιθουανία δεν θεωρούν ότι η, γλώσσα, η γνώση της επίσημης γλώσσας είναι απαραίτητα ένα προσόν ε, για την ε, αγορά εργασίας. Θεωρεί ε, ο κ. Στομασεύσκη ότι και στην Πολωνία πλήττονται οι μειονότητες. Η κυρία Ζαμπόρκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ανέφερα στη συζήτηση και εκτίμησα ιδιαίτερα το γεγονός ότι η κυρία Χάνιμπολ προσπάθησε να βρει συνένεση σε όλο το πολιτικό φάσμα. Παρ' όλα αυτά αποφάσισα να απόσχω στη ψηφοφορία διότι θεωρώ ότι η έκθεση αυτή υπερβαίνει ε, και περνά στα αρμοδιότητες των κρατών μελών. Παραδείγματο χάρη, χαιρετίζει του στόχους της Βαρκελόνη. Αλλά οι στόχοι της Βαρκελόνη κατέληξαν σε, ένα, σε αποτυχία. Και αυτό γιατί προσπαθήσαμε να ε, περάσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο πράγματα τα οποία ήταν αρμοδιότητα των κρατών μελών. Θα πρέπει να αποφασίσουμε ε, τι θέλουμε. Δεν είναι όμως θέμα μόνο αριθμητικών στοιχείων αλλά και ποιότητας. Ε, η κάθε χώρα όμως πρέπει να το αποφασίζει ατομικώς λυπάμαι που δεν μπόρεσα να υποστηρίξω τη συγκεκριμένη έκθεση, αλλά είναι κατά των αρχών μου σε βασικές ουσιώδεις πτυχές. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στην ε, Συμφωνία Λευτική Σύμπραξη μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαυριτανίας. Συγγνώμη κυρία Πρόεδρε. Ήθελα να μιλήσω και για το σημείο αυτό. Μπορώ. Σας έχω εγγράψει τον κατάλογο για άλλες ε, εκθέσεις. Δεν πειράζει, πέστε μας. Κυρία Πρόεδρε, τα πρώτα παιδικά χρόνια σαφώς έχουν σημαντική επιρροή για την ανάπτυξη ενός παιδιού και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να επενδύσουμε λοιπόν στην παιδεία και σαφώς ε, ε βοηθούμε ιδιαίτερα τον καθένα να αναπτυχθεί καταλήλως. Η φυσική υποστήριξη είναι ε, ο οικογενειακός πυρήνας, διότι οι γονείς είναι η πρώτη παιδαγωγή των παιδιών τους. Δεν θα πρέπει λοιπόν να αναφερθούμε εδώ και στο στοιχείο αυτό. Να λέμε για παράδειγμα ότι αν οι γονείς δεν φροντίζουν τα παιδιά τους ε, στα πρώτα παιδικά τους χρόνια θα πρέπει ε, με κάποιο τρόπο να τιμωρούνται. Πρόκειται για ένα στοιχείο το οποίο είναι σημαντικό και θεωρώ ότι θα μπορέσει να βελτιώσει την κατάσταση των οικογενειών στα κράτη-μέλη. Περνάμε τώρα στην ελευτική σύμπραξη μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαυρτανίας, ο κύριος Χάναν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλοί υποστηρίζουν ότι τα ψάρια δεν γνωρίζουν σύνορα. Δεν σας λέω και κάτι καινοφανές. Νομίζω ότι είναι γνωστό ότι σπάσει αυτό. Κι όμως περιφερειακή δικαιοδοσία και τα δικαιώματα ιδιοκτησία είναι αυτά τα οποία καθορίζουν τα δυνατότητε διατήρηση ελευτικών αποθυμάτων. Δείτε ποιοι καταφέρουν να τα διατηρούν. Τα νησιά Φόκλαντ, η Ισλανδία, η Νέα Ζηλανδία. Όλοι κατάφεραν να το κάνουν αυτό δίνοντα στου ε, κυβερνήτε των ε, σκαφών μια αίσθηση ιδιοκτησία και έτσι μεταχειρίζονται και τα ψάρια ω ε, ανανεώσιμε πηγέ. Αυτό λέει άλλωστε και ο Αριστοτέλη. Αν δεν σου ανήκει κάτι, δεν σε ενδιαφέρει τα αλλιευτικά αποθέματα παρόλα αυτά ε, τα αντιμετωπίζουμε ως κάτι στο οποίο έχει ο καθένας πρόσβαση, γι' αυτό και έχουμε και τις φυσικές καταστροφές που αντιμετωπίζουμε. Τα τελευταία χρόνια διαπιστώσαμε ότι το σκουμπρί ε, μεταφέρεται από τα ευρωπαϊκά ύδατα αλλιεύσης ε, στην Ισλανδία. Δυστυχώς αυτό το κάνει η διοκτησία της Ισλανδίας. Κακή τύχη δική μας, καλή τύχη για αυτούς, μπορεί να αντιστραφούν τα πράγματα σε κάποια χρόνια, αλλά προ το παρόν έτσι έχουν τα πράγματα. Προς το παρόν η καλύτερη η διασφάλιση ότι θα έχουμε τα αλλιευτικά αποθέματα που χρειαζόμαστε είναι να υπάρχει κατάλληλη αναγνώριση της ιδιοκτησίας στα θαλάσσια ύδατα. Περνάμε τώρα στις δημόσιες συμβάσεις. Ο κύριος, κύριε Μικολάσιτς, εδώ σας έχω εγγεγραμμένο στο κατάλογο για τις δημόσιες προμήθειες. Όχι, κυρία Πρόεδρε, ήθελα το λόγο και για ε, το Small Business Act. Για το συγκεκριμένο θέμα δεν ήθελα να μιλήσω. Ωραία. Να περάσουμε λοιπόν στην κρίση στον τομέα της Ευρωπαϊκής Αλίας λόγω της αύξησης των τιμών του πετρελαίου. Ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η τιμή του πετρελαίου δεν είναι η μοναδική αιτία για την κρίση στην ε, Αλία, διότι στο κάτω της γραφής η τιμή του πετρελαίου επιδοτείται <clears throat> για την ε, Αλία. Χρειάζεται βέβαια ενίσχυση των ψαράδων ώστε να εργαστούν με τρόπο βιώσιμο και αηφόρο. Και μόνη η επιδότηση του, της τιμής του πετρελαίου δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα χρειάζεται να βρεθούν και άλλες καινοτόμες λύσεις από τις χώρες μέλη. Ευχαριστώ κυρία Μπουλμπάου Μπαραντίκα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω και εγώ τα συλληπιτήριά μου στους κατοίκους της Λόρκα, της Μούρθια, της Ισπανίας, τα οχτώ θύματα, τις οικογένειές τους και τα 250 άτομα που τραυματίστηκαν από το χθεσινό σεισμό. Υπερψήφισα το κοινό ψήφισμα και όχι το ψήφισμα της πολιτικής ομάδα ομάδας λόγω της δύσκολης κατάστασης που βιώνει ο τομέας ο οποίος ε, πλήχθηκε έτη περαιτέρω λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου. Η αύξηση από τα 30.000 στα 60.000 ευρώ μέσα σε της επιδότησης μέσα σε τρία χρόνια μπορεί να βοηθήσει τον κλάδο σε αυτή την ε, συγκυρία και μάλιστα δεν χρειάζεται και καμία αύξηση στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δοθεί αυτή η επιπλέον επιδότηση. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ε, ε, συνθήκες και να μην στρεβλώσουμε τον ανταγωνισμό μεταξύ κρατών μελών. Θα πρέπει να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα για να μπορούν οι αλληλείς να χρησιμοποιούν καλύτερα τους ε, τα καύσιμα και να δοθούν νέε δυνατότητε στον ελευθερικό τομέα. Ευχαριστώ κύριο Σκέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, με μεγάλη χαρά υποστήριξα αυτές τις συστάσεις διότι η αλληλεία όπως και η γεωργία είναι κάτι το τελείως ιδιαίτερο, εξαρτάται από τον καιρό, παραδείγματος χάρη, παραδείγματος χάρη και ή υφίσταται τις ποσοστώσεις που βασίζονται στα αποθέματα. Τελικά η υφίσταται τις ποσοστώσεις που βασίζονται στα αποθέματα. Τελικά η Ένωση θα έπρεπε να καταλήξει να έχει μεγαλύτερη επάρκεια για να μην πω αυτάρκεια. Αυτό βέβαια θα σήμαινε και εξερεύνηση αλλιευτικών περιοχών που δεν έχουν ακόμη εξερευνηθεί αν μπορέσουμε να αυξήσουμε την προμήθεια θα επηρεάσουμε τις τιμές και φυσικά έτσι θα μειώσουμε την εξάρτησή μας από μη δημοκρατικά καθεστώτα. Ευχαριστούμε και τώρα το Small Business Act. Ο κύριος Ρόδα δεν φαίνεται να είναι εδώ. Δεύτερος ο κύριος Μικολάσικ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ ότι το Small Business Act πρέπει να επανεξετάζεται περιοδικά και από τα κράτη-μέλη και σε ενωσιακό επίπεδο διότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχογοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και δίνουν πάνω από 100 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Τα πράγματα δείχνουν ότι σε περιφερειακό επίπεδο η χρηματική στήριξη για την καινοτομία ή για την ίδρυση μιας μικρομεσαίας επιχειρήσης δεν είναι επαρκής. Και μελέτες δείχνουν ότι μέσω μεσολαβητικών τραπεζών 75% Thank you, uh, χορηγείται μόνο των δανείων που εγκρίνονται. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ας μιλήσω και εγώ λίγο για αυτό το θέμα. Υποστηρίζουμε την κύρια ιδέα της έκθεσης για οποιαδήποτε στήριξη των ΜΜΕ και στην Ιρλανδική και στην Ευρωπαϊκή οικονομία. Δεν βλέπουμε όμως γιατί χρειάζεται να αναφερθεί εδώ η CCCTB που λέμε. Στη Γερμανία δεν το δέχονται αυτό το CCCTB που λέμε. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζεται αυτό το CCCTB που λέμε και άλλες που δεν χρειάζεται. Συμφωνώ λοιπόν να στηριχθούν οι ΜΜΕ αλλά όχι το CCCTB. Δεν θέλαμε να καταψηφίσουμε το σύνολο της έκθεσης αλλά έπρεπε να σας πω τη λεπτομέρεια αυτή για το CCCTB. Κύριε Μίτσελ, θα ήθελα να σας θέσω εγώ μια ερώτηση. Μπορείτε να μας πείτε τι είναι αυτά τα CCCTB που μας λέτε. Χαίρομαι που το ρωτήσατε διότι ε, φάνηκε σαν να μιλάω λιθουανικά. CCCTB είναι κοινή φορολογική ε, βάση επιχειρήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Κοινή φορολογική βάση επιχειρήσεων. Είμαι βέβαιη ότι θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα οι επισκέπτες μας τα θεωρία, το γεγονός ότι γνωρίζουν πλέον γιατί ακριβώς μιλάμε. I was just about to ask whether some... Ήθελα να ρωτήσω αν κάτι μπορεί να είναι ιδεολογία ακριβώς επειδή δεν βρίσκεται στην Ιρλανδία. Δεν είναι ερώτηση για το πώς έχουν τα πράγματα στην Ιρλανδία. Δεν είναι αυτό το θέμα. Εμεί είμαστε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε παρουσιάσει τι απόψει μα και δεν θα μα υπαγορεύσει τι να κάνουμε κανένα εκπρόσωπο, κανό κράτου μέλου. Δεν υποχρεώμαστε στη χώρα αυτή να κάνουμε ό,τι κάνουν και άλλε χώρε μέλη. Ο καθένα στέλνει του ευρωβουλευτέ του εδώ για να παρουσιάσει τι απόψει του. Και η άποψή μα είναι ότι στην περίπτωση αυτή τη κοινή φορολογική ε, βάση, η οποία αποφασίστηκε το Βερολίνο, στο Βερολίνο και είναι ε, ανοησία που επινόησε κάποιον, δεν μα βοηθά δρά κατά ημών και θα πρέπει να μην υποκύψουμε σε οποιαδήποτε βούληση του καθενός. Εδώ είμαστε στη διαδικασία επεξήγησης ψήφων. Σας παρακαλώ ηρεμία. Ο κύριος Τάκουλα. Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά την κοινή φορολογική βάση, είναι πολύ καλό το ερώτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τα 27 κράτη-μέλη διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Έχουν διαφορετικές δομές ε, και διαφορετική λειτουργία. Αλλά επειδή έχουμε νέα αγορά, είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πράγματι θα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έχουν κατάλληλου κανόνε ανταγωνισμού. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή, γι' αυτό ακριβώς και διεξάγουμε και μία έρευνα και εξετάζουμε τι γίνεται με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η Φιλανδία είναι μια χώρα στην οποία οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν καμία σχέση με τον πυρήνα της ενιαίας αγοράς. Έχουν ε, αλλάξει πολύ σημαντικά οι τιμές των προϊόντων μας και χρειαζόμαστε ένα αντιστάθμισμα με διαφορετικό τρόπο, είτε μέσω μιας ευρωπαϊκής φορολόγησης, είτε μέσω κάποιου άλλου τρόπου, ώστε να μπορεί να είναι πιο ισότιμος ο ανταγωνισμός. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ετοιμάστηκε μια τέτοια έκθεση και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι ακόμα και οι πιο απομακρυσμένες, οι πιο βόρειες περιοχές και οι επιχειρήσεις τους θα έχουν ίσες δυνατότητες ανταγωνισμού με άλλες περιοχές του κόσμου. Κύριο Κέλλη. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τα όσα είπε ο Γι Μίτσελ για, την, ε, για το CCTP και θα ήθελα να επικεντρωθώ και σε ένα διαφορετικό σημείο. Ήταν αξιοσημείωτο το γεγονό ότι χρειάστηκε προφορική τροπολογία για να τεθεί το θέμα της παραποίηση για την πρόταση αυτή. Τα παραποιημένα προϊόντα είναι ιδιαίτερα επιζήμια για τις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη και δεν επισημαίνεται το θέμα επαρκώς. οι κυβερνήσεις των χωρών που παράγουν παραποιημένα προϊόντα διευκολύνουν ε, την εισαγωγή στην Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να, κατανομήσουμε αυτές τις χώρες, να κατανομάσουμε αυτές τις χώρες και να αναλάβουμε και δράση διότι έχουν πολύ σημαντικές συνέπειες για ε, ε, καθόλου ανώμιμες επιχειρήσεις και νομίζω ότι ήγηκε και η ώρα να δράσουμε πλέον. Έκθεση Μακής για την καινοτομία. Ο κύριος Πίλαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η αποτελεσματικότητα και ε, η ανταγωνιστικότητα είναι οι καλύτερες μέθοδοι για την ανάπτυξη και για να τις πετύχουμε χρειάζεται συγκεκριμένη και συνδυασμένη δράση υπέρ της καινοτομίας. Παραδείγματος χάρη να επιτρέψουμε στους εργαζομένους να υποβάλουν προτάσεις για την αποτελεσματικότερη εργασία των. Είμαι σίγουρος ότι οι πολίτες μας θέλουν παραδείγματο χάρη να χρησιμοποιούνται τελευταίας λέξης τεχνολογίες όπως το iPhone, το iPhone. Ξέρουμε όμως ότι οι ακαδημαϊκοί κύκλοι και οι επιχειρήσεις πρέπει να συνδυαστούν για να γίνει κάτι τέτοιο. Και άρα χρειάζεται καλύτερη συνεννόηση και με τις τοπικές αρχές για να παραμείνει ο πλούτος μας μέσα στην Ευρώπη. Α, αυτό άκουσα. Ο κύριο Γιάρ, δεν είχαμε δυνατότητα στη συζήτηση παρόλο που ήμουν παρόν να παρέμβω. Ωστόσο θα συμφωνήσω με τους αγορητές εκείνους που τόνισαν ότι η έρευνα και η καινοτομία πρέπει να διεξάγεται και στον αγροτικό τομέα. Η αγροτική οικονομία δεν είναι ξεπερασμένη. Είναι σύγχρονη οικονομία και έχει ανάγκη από την καινοτομία. Τρεις είναι οι μεγάλες προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Πρώτα η διασφάλιση της ανθρώπινης διατροφής. Δεύτερο η παραγωγή και προστασία του περιβάλλοντος ταυτόχρονα και τρίτο η παραγωγή ενέργειας. Αυτά, αυτοί οι στόχοι που εν μέρει αποκλίνουν χρειάζονται επιστημονική θεμελίωση και παρακολούθηση και σήμερα και στο μέλλον. Σιόκρε. Κυρία Πρόεδρε, εγώ υπερψήφισα την έκθεση για την Ένωση για την Καινοτομία αλλά νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι να στηρίξουμε την καινοτομία ιδίως στις ΜΜΕ και ε ιδίως δε στις νεότερες χώρες μέλη όπου σημειώνονται απαράδεκτες καθυστερήσεις στον τομέα αυτών Γιατί αν θέλουμε να παραμείνει ανταγωνιστική η ευρωπαϊκή οικονομία σε σύγκριση με άλλες μεγάλε οικονομίες πρέπει να στηρίξουμε τι ΜΜΕ. Διότι αυτό δείχνει η έρευνα, αυτό δείχνει. Ότι τρεις από τις τέσσερις εφαρμογές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να για να χρησιμοποιήσουν τι νέε τεχνολογίε, δεν χρηματοδοτούνται επαρκώ ή απορρίπτονται τα σχέδια αυτά. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάτι παραπάνω για να πιστούν τα κράτη-μέλη να υποστηρίξουν τι μικρομεσαίες επιχειρήσει και στον τομέα αυτών. χωρί τέτοια στήριξη δεν θα μπορέσουν να τα καταφέρουν από μόνε του μπροστά στην αυξανόμενο ανταγωνισμό διεθνώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Κούτκι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ υπερψήφισα την ενδιαφέρουσα αυτήν έκθεση για την μετατροπή της Ευρώπης σε έναν κόσμο μετά την κρίση. Ελπίζω η διαρροή εγκεφάλων να μειωθεί και να διασφαλιστεί βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό θα γίνει μόνο αν δώσουμε περισσότερα χρήματα στην καινοτομία και την έρευνα. πρέπει να καθοριστούν κατώτατα όρια στους προϋπολογισμούς μας για την έρευνα και την ανάπτυξη και την καινοτομία. Δεν πρέπει να τίθενται όρια και περικοπές στη χρηματοδότησή τους. Η κυρία Εκ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Γνωρίζουμε ότι η καινοτομία είναι εξαιρετικά σημαντική για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Παρά τα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μια συνολική ρύθμιση για την διαχείριση της καινοτομίας. Έχουμε τώρα την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οποία μιλεί για μια ένωση της καινοτομίας. Όμως πρέπει να εξασφαλίσουμε μια απλούστευση των κανόνων, μείωση της γραφειοκρατίας. Κάθε ερευνητής, κάθε πρόσωπο που ασχολείται στη βιομηχανία, κάθε μικρή επιχείρηση θα πρέπει να γνωρίζει ότι εάν θέλει να χρησιμοποιήσει, αν θέλει να λάβει δηλαδή δάνεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να το κάνει χωρίς υπερβολική γραφειοκρατία. Διότι τώρα αυτό είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για όλους. Επίσης να ενισχύουμε σημαντικότερα έργα και όχι μονάχα ε, πάρα πάρα πολύ μικρά. Η σύμβαση του, του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι συνθήκες εργασίας ποικίλουν και καμιά φορά είναι εξαιρετικά αρνητικές. Στην Ευρώπη έχουμε πολλούς αλλοδαπούς εργαζόμενους που έρχονται από τρίτες χώρες συχνά δεν έχουν χαρτιά εργάζονται υπό δυσχερείς συνθήκες και είναι εκτεθειμένοι στις ιδιοτροπίες των εργοδοτών πρέπει να φροντίσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων αυτών να είναι εξασφαλισμένα. Γιατί συχνά οι συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται μοιάζουν με συνθήκες σκλαβιάς. Με κακή μεταχείριση, καμιά φορά και με γενετήσεις καταχρήσεις που δεν τολμούν να τις καταγγείλουν γιατί φοβούνται μη χάσουν τη δουλειά τους. Ιδίω λοιπόν αναφέρομαι τώρα σε οικιακές βοηθούς που η προστασία τους θα πρέπει να είναι από τις πιο σημαντικές προτεραιότητες για τη στρατηγική του 2020. Ο κ. Γιάρ, για την απασχόληση σε ιδιωτικά, σε ιδιωτικά σπίτια, σε κατοικίες, οι απασχολούμενοι, οι απασχολούμενες σε αυτόν τον τομέα έχουν βεβαίως, και κυρίως για γυναίκες, έχουν βεβαίως απέτηση ορθής μεταχείρισης. Στον τομέα αυτό σημειώνονται πολλές αδικίες και πράγματα πραγματικά απίστευτα. Να μην λησμονήσουμε όμως και τη γραφειοκρατική επιβάρυνση. Για παράδειγμα στη Γερμανία τα πράγματα έχουν έτσι ώστε όταν προσλαμβάνεται κανείς στον ιδιωτικό τομέα είναι υποχρεωμένος να ζητήσει την βοήθεια φόρο τεχνικού διότι είναι πάρα πολύ περίπλοκες οι γραφειοκρατικές διατυπώσεις και οι φορολογικές. Αυτά όλα χρειάζονται ιδιαίτερη προσπάθεια και επένδυση. Όποιος λοιπόν θέλει να αποφύγει αυτά, εν τέλει πληρώνει ε, τα χρήματα αυτά μέτρητής που τους ζητούν δηλαδή, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση μιας παραοικονομίας. Τώρα, αντίσταση στα αντιβιωτικά. Πάλι ο κύριος Κυρία Πρόεδρε, θα μπορούσα να παραμείνω και όρθιος βέβαια και να μην καθίσω στο μεταξύ. Εγώ είμαι βέβαια εξ επαγγέλματος Γεωργός για το θέμα αυτό έχω λοιπόν πολλά να πω. Η αξίωσή μας θα πρέπει να είναι η χρήση των ιδιωτικών, κυρίως στα ζώα να μειωθεί. Low as possible θα πρέπει να είναι η βασική γραμμή της δράσεώς μας. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης. Τι συμβαίνει δηλαδή στις χώρες μέλη. Όλες οι χώρες μέλη θα πρέπει να συμμετάσχουν στην ανάλυση αυτή. Τρίτο, χρειαζόμαστε περαιτέρω επιστημονικές έρευνες για την ανάλυση των κινδύνων και για να μπορέσουμε έτσι να αντιμετωπίσουμε ορθά τους κινδύνους. Αυτό που δεν χρειαζόμαστε είναι η ιδεολειψία, διότι η ιδεολειψία δεν μπορεί να αντικαταστήσει την επιστημονική θεώρηση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και για την υπομονή σας. Έκθεση σόκο για την πολιτιστική διάσταση της Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Υπηρεσίας. Ο κύριος Ρέπο. Υποστηρίζω βέβαια την έκθεση αυτή. Είμαστε ένας οικονομικός γίγαντας εμείς στην Ευρώπη αλλά είμαστε και πολιτιστικός γίγαντας και σε ό,τι αφορά την πολιτιστική πολυμορφία η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια μεγάλη περιοχή του κόσμου η οποία έχει ανάγκη από διπλωματική εκπροσώπηση. Όλοι έχουν δικαίωμα σε πολιτιστικές υπηρεσίες, έτσι το βλέπουμε εμείς. Και η πολιτιστική πολιτική είναι και τρόπος για να διατηρούμε επαφή με άλλες χώρες με τις οποίες έχουμε ούτως ή άλλως εμπορικές και άλλες επαφές. Γι' αυτό χρειάζεται ενίσχυση των σχέσεών μας και κυρίως με βορειοαφρικανικές χώρες οι οποίες προχωρούν τώρα στη δημιουργία δημοκρατικών κοινωνιών. Θα θέλαμε οι επαφές αυτές να έχουν πάντα σχέση και με τον πολιτισμό και όχι μόνο με την κοινωνική ευθύνη. Και θα πρέπει τα πολιτιστικά να περιληφθούν με τρόπο διαρθρωτικό στην εξωτερική πολιτική της Ένωσης. Ο κύριος ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν πολιτιστικές διαφορές μεταξύ των, αλλά υπάρχει και ένα σήμα κατατεθέν πλέον ε, ανά τον κόσμο που τους επιτρέπει να ε, προσελκύουν και πολλούς πολίτες από άλλες χώρες του κόσμου. Η οικονομική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να ενισχυθεί ακριβώς δίνοντας τη δέουσα σημασία στις πολιτιστικές αξίες η πολιτιστική βιομηχανία ε, είναι αυτή η βιομηχανία η οποία δίνει τη δυνατότητα ε, στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ενώ στις χώρες στις οποίες υπάρχει λογοκρισία ακριβώς καταπιέζονται οι πολίτες της. Μέσω του διαδικτύου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υποστηρίζει τους πολίτες τρίτων χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο και να ε, μπορέσουν να το συνειδητοποιήσουν αυτό οι πολίτες. Θα πρέπει να υπάρχει ανάπτυξη της κινητικότητας για τους νέους στη διάρκεια της ε, ανάπτυξης και της μόρφωσής τους. Είμαι υπέρ της, ε, του πολιτισμού γι' αυτό και περιψήφισα αυτή την έκθεση. Ο κύριος... Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις στην έκθεση οι οποίες είναι πολύ εύστοχες και πολύ επίκαιρες. Για παράδειγμα λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δράσει παγκοσμίω υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης, της ελευθερίας της σκέψης και ε, της ελευθερίας των ε, τηλεοπτικών και οπτικοακουστικών μέσων. Υπάρχει επίσης και μία ε, όθηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προάγει την ελευθερία στο διαδίκτυο, η οποία ελευθερία είναι όλο και περισσότερο σε κίνδυνο. Θυμόμαστε λοιπόν ότι αυτές είναι θεμελιώδεις αξίες για μας τους Ευρωπαίους, αλλά συνειδητοποιούμε ταυτόχρονος ότι πολύ συχνά αναφερόμαστε σε αυτές τις θεμελιώδεις αξίες ε, και στην προαγωγή του στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά ξεχνούμε ότι παραβιάζονται ακόμα και σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε. Ως παράδειγμα σας δίνω αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Πολωνία με δημοσιογράφεις οι οποίοι ε, αρθρογραφούν κατά της ε, κυβέρνησης. Οι δημοσιογράφοι αυτοί απολύονται. Αυτό συνέβη με το δεύτερο έντυπο το οποίο είναι... Ε, το Ο κύριος Τάκουλα. Κυρία Πρόεδρε, είναι πάρα πολύ σημαντικό η πολιτιστική διάσταση να συμπεριλαμβάνεται στις συζητήσεις μας εξωτερικής πολιτικής. Διότι τώρα που συμβαίνουν τόσο πολλές διαταραχές στη Μέση Ανατολή, παρατηρούμε ότι το έχουμε ξεχάσει για δεκαετίες μάλιστα παραδείγματος χάρη στις σχέσεις μας με τη Συρία από το 1963 αρχίζουν να διώκουν κόσμο χωρίς δίκη να φυλακίζουν κόσμο χωρίς δίκη και εμείς βλέπουμε μόνο τα εμπορικά στοιχεία των σχέσεών μας και τα οικονομικά όπως είπε και η συνάδελφος Ρέπο όμως, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι βασικό στοιχείο της πολιτιστικής διάστασης. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία. Αυτά πρέπει να εξάγουμε στην ε, πολιτική μας και όχι μόνο τα οικονομικά. Ευχαριστούμε Κούσκι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ υπερψήφισα την ενδιαφέρουσα αυτή έκθεση για την πολιτιστική διάσταση των ευρωπαϊκών εξωτερικών δράσεων. Δεν θα μπορούσα να δεχτώ όσους λένε ότι προωθούμε τη δημοκρατία και την ελεύθερη πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης παγκοσμίω, αλλά, αλλά αγνοώντας τι συμβαίνει μέσα στην Ένωση. Στην Πολωνία παραδείγματος χάρη από τότε που πήρε την εξουσία ο συνασπισμός διώκονται δημοσιογράφοι που επικρίνουν την κυβέρνηση όπως ο Γιάτσεκ Σομπάλα, η κυρία Γκάργκας και άλλοι έχουν απολυθεί άλλοι σε άλλους απαγορεύτηκε το δικαίωμα εργασίας στα μέσα ενημέρωσης. Αυτά όλα είναι σχρά. Ευχαριστούμε. Να με προσέξει ο κύριος Τάκουλας. Έχουμε έρθει στην τελευταία έκθεση Σάντσες Σμιτ και το Σαράγεβο σαν πολιτιστική πρωτεύουσα. Ζητήσατε επεξήγηση και για τις δύο τελευταίες αυτές εκθέσεις. Έχετε τον λόγο ότι η μία μετά την άλλη να τις κάνετε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτον, για τη Σάντσις Σμιθ. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε την αξία του πολιτισμού και των δημιουργικών βιομηχανιών ή των βιομηχανιών δημιουργίας. Το 2,6% του ΑΕΠ μας από αυτές προέρχεται και απασχολεί το 3,1% του δυναμικού μας. Τις τελευταίες δεκαετίες αναπτυσσόταν συνεχώς. Αλλά η πολιτιστική διάσταση σημαίνει επίσης ότι δεν υπάρχουν μόνο τα οικονομικά και η ανάπτυξη, υπάρχει και η ανάπτυξη και εξέλιξη των ανθρωπίνων όντων. Δεν πρέπει λοιπόν να τα μετράμε όλα μόνο με το ΑΕΠ, αλλά να καταλαβαίνουμε ότι το πρόσωπο δεν έχει σαν σκοπό μόνο να παράγει και να καταναλώνει. Και αυτό όμως απαιτούνται ορισμένοι όροι και πρέπει να το καταλάβουμε και εμείς ως ευρωβουλευτές. Ιδιαίτερα συχνά περιορίζουμε την Ένωση μόνο σε αυτά τα στοιχεία τα οικονομικά. Τώρα για το Σαράγεβο ως πολιτιστική πρωτεύουσα το 2014 θα ήθελα να πω ότι είναι μια ιδέα που προήλθε με μεγάλη συνένεση από την Πολιτιστική Επιτροπή γιατί πρόκειται για εκατοστή επέτειο της αρχής του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και θέλουμε να δείξουμε το 2014 ότι ότι λέγω θέλουμε να εγγενιαστεί τότε ένας αιώνας ειρήνης ιδιαίτερα στα Βαλικάνια Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Εδώ έληξαν και οι επεξηγήσεις ψήφου. Στις 3 θα ξαναρχίσει η σύνοδος. Σας ευχαριστώ.